Okej. Okay. Eh, god eftermiddag allihopa. Eh, ja, eh. Καλώς ορίσατε. Θα μπορούσατε να φορέσετε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω σε ειδικά. Έτοιμοι. som är då Έχουμε φτάσει εσείς στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης, την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Έχουμε εδώ μαζί μας την κυρία Βιρτζίνια Λάγκπακ, η οποία θα μας παρουσιάσει αυτή την ετήσια έκθεση και κατόπιν θα έχουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Παρακαλώ κυρία Λάγκπακ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πρόσφατη επίσκεψη της Επιτροπής ε, Γυναικών ήταν ιδιαίτερη για μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Αντιπροσωπεία και τον Πρόεδρο για την επίσκεψη και για τις ε, συζητήσεις. Ε, ακόμα ε, είμαστε σε διάλογο με όσους συμμετείχαν και για μας υπήρξε ορόσημο αυτή η στιγμή διότι μπορέσαμε να δούμε τι κάνουμε και ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η επίσκεψή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τώρα την ετήσια έκθεση. Από ό,τι βλέπω την έχετε ήδη λάβει. Ε, έχουμε τυπώσει μόνο το πρώτο τμήμα για την ε, ε, διάσκεψη και τώρα ζητήσαμε να σταλεί και το δεύτερο, ειδικά για σας για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Ε, το βασικό είναι ότι υπάρχουν δύο εκθέσεις, όπως κάνουν οι περισσότεροι αποκεντρωμένοι οργανισμοί. Η μία έκθεση ενδιαφέρεται περισσότερο για τα θέματα ισότητας φίλου και αυτή είναι η ετήσια έκθεση την οποία δημοσιεύουμε. Και η δεύτερη έκθεση είναι αυτή που έχουμε αποστείλει στο Κοινοβούλιο μόνο ηλεκτρονικά και είναι μια πιο διοικητική φύσεως έκθεση που αφορά τις δραστηριότητές μας και φυσικά έχει σχέση και με τη διαδικασία απαλλαγή ε, όταν εξετάζει το Κοινοβούλιο πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια και κατά πόσον επετέφθησαν οι στόχοι. η μία εξετάζει τα πράγματα απλώς από πλευράς φίλου ε, είναι πιο σαφ... και η άλλη είναι πιο διεξοδική και δεν την εκτυπώνουμε, την έχουμε μόνο διαδικτυακά. Τώρα, πριν ξεκινήσω την παρουσίαση, ίσως ε, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι το 2012 ήταν η τελευταία χρονιά του πρώτου τμήματος ε, του προγράμματος εργασίας μέχρι την ε, έγκριση δηλαδή των πρώτων τριών ετών. Το 2009 εγκρίθηκε το πρώτο μεσοπρόθεσμα τριετές πρόγραμμα και έχουμε το διάστημα 2009-2012 και θα δείτε ότι υπάρχει και ένας πίνακας στον οποίο γίνεται ένας έλεγχος όλων των αποτελεσμάτων και εκεί μπορείτε να δείτε και την συγκεκριμένη παρακολούθηση των θεμάτων αυτά τα οποία προσπαθήσαμε να επιτύχουμε και ποιους θεωρούμε στόχους εν γέννη, θεωρούμε ότι τα έχουμε όλα υλοποίησει. Στην επόμενη διαφάνεια ε, δεν έχω και πολλά να πω. Μας επισκέφθηκε ήδη η Επιτροπή Γυναικών. Στη διάρκεια του περασμένου έτους οριστικοποίησαμε όλες τις διαδικασίες ε, για τη μόνιμη έδρα μας. Και όπως βλέπετε, εδώ έχουμε την έδρα μας και μοιραζόμαστε την έδρα αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, προσπαθούμε να δούμε τι συνέργειες έχουμε, κατά πόσον υπάρχει αποτελεσματικότητα, αλλά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το θέμα αυτό, για το γεγονός ότι συστεγαζόμαστε. για τη σύσταση του οργανισμού ε, υπογράψαμε πέρσι και μια συμφωνία για την έδρα και αυτό αποτελεί προϋπόθεση μεταξύ της χώρας υποδοχής και του οργανισμού για όλους τους ε, αποκεντρωμένους οργανισμούς. Ολοκληρώθηκε και αυτό και τώρα στην επόμενη διαφάνεια Uh, έχουμε τα στοιχεία για το προσωπικό. Έχουμε 19 εθνικότητες, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 39 ετών, ε, έχουμε 51 ε, άτομα στο προσωπικό και συμβασιούχους ε, και εθνικούς εμπειρογνώμονες και εκπαιδευόμενους κλπ. Ε, αν δείτε τώρα την ε, διαφάνεια για την εξέλιξη και τις προβλέψεις μας, θα δείτε πώς σκοπεύουμε να ε, κάνουμε προσλήψεις και τι έγινε με το προσωπικό μας. Και πάλι κάναμε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες από το 2010 και τούδε να τηρήσουμε το, το οργανόγραμμα και είχαμε άλλους δύο συμβασιούχους το 2010. Φτάσαμε λοιπόν στο 50% ε, το 2012 και μετά όσα προβλέπουμε και από το σχέδιο προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε 30 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και τους υπόλοιπους ε, ε, με άλλες συμβάσεις. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε στον προπολογισμό και είδαμε τι εκκρεμεί, τι δεν χρησιμοποιήσαμε και θα είναι πλεόνασμα για του χρόνου και θα ήθελα να σας δείξω λίγο και το γράφημα που έχουμε στην επόμενη διαφάνεια, όπως θα δείτε στο ε, διάγραμμα αυτό έχουμε πόσο αποτελεσματικός είναι ο προϋπολογισμός και πόσο γρήγορα γίνεται ο προγραμματισμός για τις δραστηριότητές μας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από αρχές του 2013 να εξετάζουμε κάποια προγράμματα, τα παρακολουθούμε στενά ώστε να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση και να προσπαθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να είναι όλα προγραμματισμένα ώστε να απορροφάται όλος ο προϋπολογισμός βάσει των δραστηριοτήτων μας. Στην επόμενη διαφάνεια, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εδώ έχουμε ε, βελτιώσεις στα ποσοστά και για τις ε, δεσμεύσεις και για τις πληρωμές. Ε, αυτά θα τα έχουμε και στην διοικητική έκθεση, αλλά θεώρησα ότι επειδή εσείς είστε η αρμόδια επιτροπή για μας, ήταν σημαντικό να σας δείξουμε πώς προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Τώρα, προμήθειες στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε λίγο πολύ τα γενικά στοιχεία, όπως έγινε και την προηγούμενη χρονιά. Καθυστέρησε πάρα πολύ η απόφαση από πλευράς μίας εκ των Προεδριών και έτσι είχαμε καθυστερημένη μελέτη ε, και γι' αυτό χρειάστηκε να μεταφερθεί στο επόμενο έτος ε, και ε, για μία μελέτη δεν υπήρχε καμία προσφορά η οποία να είναι αποδεκτή, επομένως χρειάστηκε να προκηρυχθεί εκ νέου ο διαγωνισμός. Περνάμε τώρα στις εργασίες μας ε, για το ότι κάνουμε για την ισότητα των φύλων. Εδώ ε, βλέπουμε πού εστιάζουμε. Στη διάρκεια του περασμένου έτους επεκτείναμε τις συζητήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθήσαμε να διευρύνουμε λίγο την ε, βία κατά των γυναικών ε, είχαμε κάποιες εκθέσεις. Στη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ε, έγινε και μία έκθεση για την προστασία των θυμάτων και τη στήριξη στα θύματα και συζητήσαμε βέλτιστες πρακτικές, ε, διάφορα εργαλεία, συλλέξαμε διάφορα στοιχεία και θα υπάρξει και μια σχετική δημοσίευση για να υποστηρίξουμε αυτές τις πρακτικές και να δείξουμε στα κράτη-μέλη πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Εδώ ε, κάτι που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ε, Γυναικών, το θέμα του ακροτηριασμού γενετικών οργάνων. Ε, το παρουσίασε και την πρόεδρος Ρέντινγκ το Μάρτιο και παρουσιάσαμε, αναπτύξαμε το σχετικό πρόγραμμα και συλλέξαμε στοιχεία και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την παρακολούθηση του θέματος αυτό και για του χρόνου. Θα δούμε τώρα τι αποτέλεσμα θα έχουμε μετά από τη διαδικασία διαβούλευσης της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ, να καθοριστούν κάποιες προτεραιότητες και μετά. Στην επόμενη διαφάνεια έχουμε τη βία βάση του φύλου και εδώ έχουμε συλλογή δεδομένων στο διοικητικό επίπεδο. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μελέτη που ολοκληρώνεται φέτος αλλά ξεκίνησε πέρσι. Εάν θέλουμε να έχουμε δείκτες, αν θέλουμε να αρχίσουμε να παρακολουθούμε και να μετρήσουμε τι γίνεται στα θέματα της βίας κατά των γυναικών, θα πρέπει να δούμε τι δεδομένα έχουμε και θέλουμε να ξέρουμε και τι ε, δεδομένα έχουμε, αξιόπιστα δεδομένα σε επίπεδο κρατών μελών. Έγινε μία σε την περασμένη εβδομάδα και με βάση αυτά θα συνεχίσουμε ε, τις εργασίες μας και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Γυναικών για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεδομένα υπάρχουν. Κατόπιν, από ό,τι βλέπετε έχουμε πάνω από 26.000 αναφορές σε διάφορες γλώσσες ε, κατά βάση τις τρεις ε, βασικές γλώσσες αλλά και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκονται ε, σε άλλες γλώσσες και έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες δημοσιεύσεις και, πόρου, και πηγές και που χρησιμοποιούνται αλλά τα καιρού έχουμε και αιτήματα από κράτη-μέλη, από πολιτικούς για συγκεκριμένα θέματα και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν είτε στη γλώσσα τους είτε σε κάποια άλλη γλώσσα για να μπορέσουν να λάβουν τις αποφάσεις τους. Εδώ, στη διαφάνεια αυτή, έχουμε αξιόπιστα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αναπτύξαμε δύο δείκτες πέρσι, τους γνωρίζετε αυτούς τους δείκτες, τέσσερις συγγνώμη νέους δείκτες, ε, οι περισσότεροι σχετίζονται με την έκθεση της Δανικής Προεδρίας για τις γυναίκες και το περιβάλλον συλλέχθησαν νέα στατιστικά στοιχεία βάσει αυτών των δικτών και κατόπιν το Συμβούλιο ενέκρινε τους νέους ε, δείκτες ε, για το φύλλο και την ε, κλιματική αλλαγή για πρώτη φορά και έχουμε και δύο νέες σειρές δεδομένων. Όλα αυτά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα, επικαιροποιείται συνεχώς, μπορείτε κάλλιστα να κάνετε μια αναζήτηση και να βρείτε τα στοιχεία που θέλετε. Και ε, θα συμπεριληφθούν και στη βάση δεδομένων <clears throat> όχι φέτος αλλά την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο υπάρχουν δύο νέες σειρές δεδομένων που προέκυψαν και πάλι από την Κυπριακή Προεδρία για την υποστήριξη των θυμάτων βίας και για τα θέματα γυναικών και περιβάλλοντος. Στην επόμενη διαφάνεια ένα παράδειγμα ε, των όσων ξεκινήσαμε τον Απρίλιο και χάρηκα ιδιαίτερα που ήταν παρόν ο πρόεδρος Επιτροπής ε, Γυναικών που ε, ήταν εκεί, συμμετείχε στη διάσκεψη ε, είναι πολύ καινούργια αυτά τα πράγματα. Ε, ξεκινούμε τις εργασίες μας. Υπάρχουν διάφορα αιτήματα από κράτη-μέλη και χρήστες ε, περισσότερο για το πώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα νέα στοιχεία. Θα δούμε και με τα κράτη-μέλη που μπορούμε να διευρύνουμε λίγο κάποιους συγκεκριμένους τομείς εργασίας. Θα πρέπει ε, για το δίκτυ ισότητας να δούμε και κάποια θέματα, τη βία για παράδειγμα ε, και κάποιες διασταυρούμενες ανισότητες, πώς θα τα εντάξουμε στη συζήτηση. Όλα αυτά όμως ε, προέκυψαν ως ένα πολύ καλό αποτέλεσμα μετά από τρία χρόνια δουλειάς. Αποτελεσματικές πολιτικές και εφαρμογή τους τώρα. Εδώ έχουμε την ε, διαδικτυακή βάση δεδομένων που βασίζεται περισσότερο στα θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και είχαμε και εκπαιδευτές, ε, ε, έγιναν και κάποια σεμινάρια, δημοσιεύσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε δύο βάσεις δεδομένων και αρκετές πηγές οι οποίες από ό,τι γνωρίζω χρησιμοποιούνται και τώρα ετοιμάζουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης για το πώς θα επικαιροποιήσουμε και θα γνωστοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία και πώς θα γνωρίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι κυβερνήσεις ότι υπάρχουν κάποιες καλές πηγές ώστε να εξοικονομούν και χρόνο και χρήμα χρησιμοποιώντας τις. Έχουμε τώρα ένα κέντρο ε, τεκμηρίωσης ε, Φιλοδοξία μας είναι να τα έχουμε όλα σε ένα σημείο, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να αναζητά παντού πού θα βρει όλα τα στοιχεία που αφορούν την ισότητα των φύλων. Θέλουμε να είναι συγχρονισμένος ο τρόπος παρουσίασης αποτελεσμάτων, ώστε να μπορεί κάποιος με ένα απλό κλικ να βρει τα στοιχεία που θέλει. Όπως βλέπετε, δεν έχω και τα γυαλιά μου, Έχουμε πάνω από 26.000 πηγές σε διάφορες γλώσσες, επικαιροποιούνται συνεχώς και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι συλλέγουμε στοιχεία και βιβλιογραφία που δεν βρίσκεται σε άλλα σημεία διαδικτυακά και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό διότι έχουμε και κάποια έγγραφα πολιτικής που χρησιμοποιούνται σε κάποια κράτη-μέλη ε, λαμβάνοντας ως παράδειγμα τι κάνουν τα άλλα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή η συνεισφορά μας εδώ. Το δοκιμάσαμε πέρσι Έχουμε και ένα ε, εικονικό δίκτυο για την ισότητα των φύλων και θέλει Θέλουμε μέσω αυτού να ε, θαρρύνουμε τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές ε, και να ανταλλάζουμε γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές. Φέτος ήδη λειτουργεί, έγιναν κάποιες συζητήσεις, θέλουμε να υποστηρίξουμε και μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στις εκλογές και φυσικά να εκλέγονται και στη συνέχεια. Έχουμε ένα ετήσιο πρόγραμμα και συζητήσαμε και με την Επιτροπή Γυναικών και είπαμε ότι θα θέλαμε και η Επιτροπή Γυναικών αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο, διότι έτσι θα έχουμε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Κατόπιν. Έχουμε και πάλι τις γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη. Είχαμε το ετήσιο ημερολόγιο, ήταν το τρίτο μας ημερολόγιο. Και Έχουμε και μία τελευταία διαφάνεια. Είμαστε στη θέση παριθμών 4 στο Facebook ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Επισκέπτονται όλο και περισσότεροι τη σελίδα μας και είμαστε πολύ περήφανοι και θεωρούμε ότι είναι και ένα από τα επιτάγματά μας για το 2012. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. για την παρουσίαση αυτή. Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο το οποίο έχουμε εγκρίνει ανάμεσα στους ε, συντονιστές και στο Ινστιτούτο αυτό για το πώς θα επικοινωνούμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το έγγραφο το οποίο περιγράφει τι θα πρέπει να κάνει το Ινστιτούτο αυτό και τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς έτσι ώστε να υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στα δύο αυτά θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δομή στην δουλειά που κάνουμε, να δούμε τι μπορεί να περιμένει ένας από τον άλλο, ποιες εμπειρίες και πρακτικές μπορούμε να ανταλλάσσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι πάρα πολύ καλό που υπάρχει δομή, που υπάρχει αυτή η συμφωνία για το πώς θα συνεργαζόμαστε. Επίσης, να πω ότι στις 13 ε, Ιουνίου συμμετείχα σε ένα συνέδριο, την ίδια ημερομηνία που ε, τέθηκε σε ισχύ η ατζέντα σας και είδα διαφορετικές πτυχές και πιστεύω ως αποτέλεσμα ότι είναι πολύ σημαντικό να διεξάγονται συγκριτικές μελέτες ε, στις χώρες εσείς έχετε ορισμένους ε, πολύ χρήσιμους δείκτες και υπάρχουν ε, κάποιες ε, χώρες όπως για παράδειγμα η Δανία, η Σουηδία και η Φιλανδία οι οποίες έχουν παρόμοια κοινωνικά συστήματα και εκεί μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις, για παράδειγμα τι λειτουργεί καλύτερα στη Δανία ή στη Σουηδία. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία Και είναι πολύ χρήσιμο να δούμε ποιες, ε, σε ποια σημεία υπερέχει κάθε χώρα, έτσι ώστε να βελτιωνόμαστε. Είναι χρήσιμο λοιπόν. Και εγώ προσωπικά θα χρησιμοποιήσω τα στοιχεία αυτά στην Σουηδία. Και αυτή τη στιγμή στη Σουηδία, κοιτάζω και τον Κέν θα μου το επιβεβαιώσει, υπάρχει μια ε, συζήτηση για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ορισμένοι λένε πως όλα είναι τέλεια, ορισμένοι λένε πως πράγματα υπάρχουν ακόμα που πρέπει να γίνουν. Αν δείτε όμως τους δείκτες θα δείτε ότι απέχουμε από το να λειτουργούν όλα υπέροχα. Είμαστε στο 74% μόνο στη Σουηδία των ε, δυνατοντήτων μας. Υπάρχει λοιπόν πολύ περιθώριο βελτίωσης. Μπορούμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σε ένα καλό εργαλείο στις ε, χώρες μας. Δεν, έχουν, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έργο μας. Ήταν πολύ επαγγελματική η παρουσίασή σας, με εξέπληξε ο τρόπος που εκθέσατε τα στοιχεία αυτά και η μεθοδολογία που ακολουθήσατε. Πιστεύω πως κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά εξηγώντας το πώς εργάζεστε, ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε, πώς συγκρίνετε τα στοιχεία που έχετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσίαση. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ομιλητές. Η κυρία Γκουρμάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι μία από τους ε, λίγους που ήταν εδώ και απόλαυσαν την παρουσίασή σας για τις εργασίες του Ινστιτούτου. Και η Edit και εγώ σας επισκεφθήκαμε και πραγματικά μας ανοίξατε την πόρτα σε ένα καινούριο κόσμο πληροφοριών. Εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω ότι έμαθα πολλά από τη δουλειά σας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι έγινε αυτή η συμφωνία με την κυβέρνηση και έγιναν και αυτές οι προπαρασκευαστικές ε, επισκέψεις εν ώψη της Λιθουανικής Προεδρίας. Να σας πω ότι οι Λιθουανοί πρέπει να είναι περήφανοι που σας έχουν στη χώρα τους. Και μου έκανε εντύπωση που μιλήσατε για τον αριθμό αυτές τις 160.000 διαφορετικές πηγές. Και μπορώ να πω ότι έχετε περισσότερες ε, πηγές και βιβλιογραφία από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαδοθεί. Και είναι επίσης πολύ καλό το ότι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σκοπό αυτό. Έχετε ένα πολύ καλό και επαγγελματικό επιτελείο και αυτό δείχνει πως με όλες τις δραστηριότητες σας είστε στην ε, ακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις. Και επίσης να πω ότι παρατήρησα ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία στις διάφορες γενιές στο Ινστιτούτο σας, στο επιτελείο σας και είναι κάτι που λείπει από πάρα πολλούς οργανισμούς. Πιστεύω πως καλό θα ήταν να έχουμε και μια παρουσίαση και εδώ για τις ε, προσεγγίσεις ε, που ακολουθούνται για να μας δώσετε και εμάς καινούργιες ιδέες εδώ τώρα για αυτά που είπατε για την κλιματική αλλαγή. Αυτά είναι νέα ευρήματα και η πράσινη οικονομία είναι κάτι που έχει συζητηθεί σχετικά πρόσφατα για το, για, ως μια πιθανή έξοδος από την κρίση. Και το θεωρώ καλή ιδέα. Τώρα, όσον αφορά την συνεκτίμηση της διάστασης του φίλου, του φίλου πιστεύω πως και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα ε, και με τον πρόεδρο που έχουμε. Και μπορώ να σας πω πως έχουμε αποκομίσει πάρα πολύ θετικές εντυπώσεις από τη δουλειά σας. Θα ήθελα Κλείνοντας να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεισφορά σας και τη δική σας και της Υπουργού σας που ήρθε σήμερα το πρωί που μας είπε για το συνέδριο το Σεπτέμβριο. Θα χαρώ πάρα πολύ να συμμετέχω στο συνέδριο αυτό. και η Επιτροπή μας θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με εσάς. Καλή τύχη λοιπόν για τις μελλοντικές σας δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε η Ζήτα, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Παρότι δεν μου έκανε τόση εντύπωση η παρουσίαση όσο έκανε στη ζήτα, διότι ήμουν μάρτυρας των προσπαθειών σας από καιρό. Και ήταν πραγματικά εκπληκτική η εξέλιξη του Ινστιτούτου σας από την αρχή μέχρι σήμερα. και δεν κάνετε μόνο καλή δουλειά, αλλά φαίνεται και καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό που με λυπεί είναι το εξής. Αρχίσατε μία μελέτη για τους ε, δίκτες του σχετικού με το φύλλο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Στρασβούργου και δυστυχώς δεν μπορούσα να συμμετέχω. Ξέρω πάντως, έμαθα ότι το συνέδριο είχε επιτυχία και η συνεισφορά του Προέδρου μας ήταν εξαιρετική. Εν πάση περιπτώσει όμως άλλο να το διαβάζεις και άλλο να είσαι εκεί. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ακούσω εσάς και θα ήθελα να μάθω Ποια θα είναι η συνέχεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να μας πείτε μερικές πληροφορίες για το τι θα γίνει με αυτόν τον δείκτη των δύο φίλων. Και επίσης θα με χαροποιούσε πολύ αν είχαμε και μια σύντομη παρουσίαση αυτών των δικτών ενδεχομένως. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Έχετε το λόγο. Ναι, όσον αφορά το δίκτυο, τους δείκτες. Εμείς ε, βεβαίως ε, με μεγάλη χαρά θα κάνουμε αυτή την παρουσίαση, όχι σήμερα, αλλά μετά το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που πραγματικά πήρε πολύ χρόνο. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος ε, δείκτης, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει. Και πρόκειται, αν θέλετε, για ένα σύστημα που μας οδήγησε σε σύνθετο δείκτη. Είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί όσα υπάρχει, αλλά το οποίο βεβαίως βασίζεται εδώ σε στοιχεία και έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήραμε όλα τα στοιχεία, όλες τις μεταβλητές, 26.000 συνολικά και προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι συγκρίσιμα και τελικά φτάσαμε σε πολύ λιγότερα στοιχεία. Όταν φτάσαμε τελικά στον τύπο που ίσχυσε για την φόρμουλα αυτού του δίκτυ, είδαμε ότι όσον αφορά τη βία δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν άδειο το τμήμα αυτό. Είχαμε λίγα στοιχεία, αλλά έλειπαν πάρα πολλά γι' αυτό και, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσουν πολύ περισσότερα στοιχεία που αφορούν το φύλλο. Επίσης υπάρχουν πολύ λίγοι δείκτες για τους άλλους τομείς που μας ε, ενδιαφέραν. Τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκουν ότι η εργασία μας είναι χρήσιμη. Άρα σήμερα μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία και δείκτες έτσι ώστε παραδείγματος χάρη να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και άλλους τομείς όπως παραδείγματος χάρη η ποιότητα της εργασίας. Σε δύο χρόνια σίγουρα όταν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας στους άλλους δείκτες, θα είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Είναι ένα μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί κανείς να διαπιστώσει τι συμβαίνει και να δει αν θέλετε κάποια τμήματα του δείκτη. δεν χρειάζεται να έχει όλη την εικόνα και τα στοιχεία είναι οπωσδήποτε συγκρίσιμα. Αυτό είναι σημαντικό για κάποιους τομείς ε, εφαρμογής. Τώρα. Κυρία Γκορμάη, χαίρομαι ιδιαίτερα που εκτιμάτε την εργασία μας, τη θεωρείτε χρήσιμη. Αναφερθήκατε σε κάποιους τομείς τους δείκτες, το gender mainstreaming. Βεβαίως εμβαθύνουμε σε αυτούς τους τομείς και θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που ιδιαίτερα ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο. Πρόεδρος. Ο κύριος Μπλάτς από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει με χαρά ότι το Ινστιτούτο συμμετέχει τακτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής σας. Έχει κατά κάποιο τρόπο ξεκινήσει ένας διάλογος και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται με πολύ τακτικό τρόπο και ρυθμό με το Ινστιτούτο. Το 2012 η κυρία Λάμπακ ήρθε σήμερα και παρουσιάζει την έκθεση δραστηριοτήτων για το 2012. Έχει γίνει λοιπόν πολύ σημαντική πρόοδος. Το Ινστιτούτο έχει επεκταθεί και το 2013 σήμερα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτό το Ινστιτούτο που είναι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία λειτουργεί με ένα πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Τώρα όσον αφορά την ποιότητα αυτής της εργασίας, εμείς επιμένουμε, η Επιτροπή επιμένει ότι η εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά ουσιαστική, πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός. Πρόκειται για μια εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη του Ινστιτούτου, την οποία πρέπει πραγματικά να συνεχίσουμε να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε. Υπάρχουν δύο θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή. Πρώτον, ο δείκτης, και εδώ χαιρετίζω πραγματικά αυτή την εργασία. Αυτός ο δείκτης παρουσιάστηκε συγγνώμη, δημοσίως πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι όμως μία δουλειά που έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια. Σήμερα απλώς παρουσιάστηκε και επισήμως ελπίζουμε στην Επιτροπή ότι αυτός ο δείκτης θα είναι χρήσιμος και θα χρησιμοποιηθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για ένα δείκτη που πρέπει να συμπληρωθεί, να ολοκληρωθεί η εργασία δηλαδή του Ινστιτούτου και αυτό που ζητάμε είναι να βελτιωθεί ο δείκτης αυτός σε δύο τομείς. Πρώτον όσον αφορά το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Όλοι γνωρίζουν εδώ ότι έχουμε πρόβλημα με την αξιοπιστία των δεδομένων στην Ευρώπη όσον αφορά αυτό το τομέα. Γι' αυτό και ζητάμε από το Ινστιτούτο να επεξεργαστεί όχι αύριο το πρωί, αλλά σιγά σιγά, μεσοπρόθεσμα, να συμπληρωθεί αυτή η έλλειψη, το κενό αν θέλετε όσον αφορά τα στοιχεία, να επεξεργαστεί τα δεδομένα που έχουν τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του δίκτυου. Η κυρία Λάμπακ είπε πολύ σωστά ότι ένας άλλος τομέας που πρέπει επίσης να συμπληρωθεί είναι η ποιότητα της εργασίας. Ο δείκτης λοιπόν είναι μια πρώτη πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία θέλει ακόμα επεξεργασία. Δεύτερος τομέας, που αν ακούσατε προσεκτικά την κυρία Λάμπακ θα το διαπιστώσετε κι εσείς, είναι η βία κατά των γυναικών. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το τομέα, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στον ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων. Και εδώ τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν είναι πλήρη σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται λοιπόν και ποσοτική αλλά και ποιοτική ε, εργασία για τον τομέα αυτό. Αυτά. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω. Διαπιστώνουμε πολύ σημαντική εργασία, πρόοδο και ζητούμε να συνεχιστεί η εργασία του Ινστιτούτου με αυτούς τους ρυθμούς. Να σας επιβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε και ότι είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε συνεχή διαβούλευση θα έλεγα. Έχουμε εξάλλου και το σχέδιο για το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2014. Είναι έτοιμο και φυσικά και θα συνεχίσουμε την επεξεργασία του δίκτυ. Σκοπός μας είναι να υποβάλουμε και ένα σχέδιο στρατηγικής για το 2014 θέτοντας προτεραιότητες. Είμαστε ένα πολύ μικρό Ινστιτούτο με πολύ μικρό προϋπολογισμό και καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ε, προτεραιότητες για τον τομέα της βίας κατά των γυναικών. Θα εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή μας στους τομείς αυτούς έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ που ήρθατε και που μας παρουσιάσατε την ετήσια έκθεσή σας. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Όπως είπατε, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία. Θα συνεχίσετε να μας επισκέπτεστε ενημερώνοντάς μας με έγγραφα, με παρουσιάσεις. Για αυτά για μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Να ξέρετε ότι η Επιτροπή μας είναι θερμός υποστηρικτής του έργου σας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ξανασυναντηθούμε πολύ σύντομα. Το φθινόπωρο θα ξανάρθετε γιατί θα μας μιλήσετε ε, πιο ολοκληρωμένα για το δίκτυ, για την ισότητα των φίλων Και σίγουρα πολύ περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι παρόντα. Εγώ τουλάχιστον θα είμαι γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο δείκτης. Ναι, πριν το ξεχάσω. Ήθελα σήμερα το πρωί να σας πω ότι η Επιτροπή Γυναικών αλλά οποιοδήποτε εδώ έχει μία πρόταση οτιδήποτε θέλετε όπως η κυρία Γκουρμάη που μόλις είπε ξέρετε ότι η Λιθουανία εμείς είμαστε στο Βίλνιους είναι η χώρα που έχει την Προεδρία. Μπορείτε λοιπόν κάλλιστα να πείτε σε μέλη των πολιτικών σας ομάδων που ανήκουν σε άλλες επιτροπές αν επισκεφθούν το Βίλνιους στο εξάμεινο της Προεδρίας να έρθουν να μας δουν. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να συναντήσουμε και μέλη του Κοινοβουλίου που δεν ανήκουν στην Επιτροπή Γυναικών, η κυρία Γκουμάη. Εγώ κάνω μια απλή πρόταση. Ο πρόεδρος μπορεί να στείλει μια επιτροπή σε όλους τους πρόεδρους επιτροπών του Κοινοβουλίου αναφερόμενος σε αυτήν την παρουσίαση που έγινε σήμερα και γραπτά να την υποβάλει σε όλους. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση. Μπορούμε να ψηφίσουμε αν θέλετε. Αλλά θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και την ε, δυνατότητα να συνεδριάσουμε εκτός Βρυξελών και φυσικά στο Βελνίος. Πρόεδρος, ναι, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν ότι εγώ, η Γραμματεία, θα... Στείλουμε αυτή την ε, επιστολή σε όλες τις επιτροπές, έτσι ώστε όταν επισκεφτούν την Λιθουανία να έρθουν να σας δουν. Συμφωνώ απολύτως, λέει ο Πρόεδρος, και θα το κάνω. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Και θα σας ξαναδούμε το φθινόπερο. Perhaps you didn't know that, but it's very... Δεν το γνωρίζετε. Αλλά είναι πολύ εύκολο να συνομιλούμε γιατί μιλάμε σουηδικά και επομένω τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Και τώρα θα μιλήσω σουηδικά και πάλι. Έχουμε φτάσει στο επόμενο σημείο, σημείο 15 στην ημερήσια διάταξη. Γυναίκες με αναπηρία. Θα δώσω καταρχώς το λόγο στην κοινή την κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η έκθεση όντως είναι πάρα πολύ σημαντική. Σκεφτείτε ότι 15% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άτομα με αναπηρία και 80% από αυτούς ζουν σε κράτη-μέλη τα οποία θεωρούνται ε, μειονεκτούντα. Η κατάσταση των γυναικών με αναπηρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπόκειται σε ε, ποικίλε διακρίσει, διακρίσει στον τομέα τη εκπαίδευση, στον κοινωνικό, τον εργασιακό, ε, στην, ε, στον τομέα τη υγεία. Οι γυναίκε αυτές πραγματικά ε, είναι θύματα δημιουργία στερεοτύπων Μίλησα με γυναίκες με αναπηρία και πραγματικά μου επιβεβαίωσαν ε, όλα αυτά και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πλέον. Προσπάθησα λοιπόν κατόπιν τούτου να γράψω μια ισορροπημένη έκθεση. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ακρόαση, πήγαν όλα καλά με την έκθεση, έτυχε καλής ε, υποδοχής υπήρξαν πάρα πολλέ επικοδομητικέ προτάσει και τροποποιήσεις τις οποίες με τα χαρά να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου και πιστεύω πως αυτό το θέμα πραγματικά μας δείχνει πόσε πολλέ διαστάσεις έχει αυτό το πρόβλημα και επίσης τότε οι γυναίκε με αναπηρία ε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ ε, δύσκολη θέση. Δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος για την ε, διάσταση των, ε, αυτή των γυναικών με αναπηρία. Να πω πάντως ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τις προτάσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκουρμάη. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη δημόσια ακρόαση νομίζω ότι έδωσε πολλά σημαντικά στοιχεία στην εισηγητριά μας και βεβαίως όταν ε, αναφερόμαστε στην κρίση αναφερόμαστε στις γυναίκες που ζουν μια σιωπηλή κρίση για τα δε άτομα με αναπηρία και τις γυναίκες με αναπηρία είναι ακόμα πιο σιωπηλή η κρίση γιατί έχουμε κράτη-μέλη που δεν έχουν καν ε, τις υποτυπώδεις ε, δομές για να τους καλύψουν. Καλό είναι λοιπόν που επισημαίνεται αυτό το πρόβλημα, διότι αν δείτε τι γίνεται με τις γυναίκες ε, με αναπηρία στην αγορά εργασίας, θα δείτε ότι είναι σχεδόν απούσες. Ε, το ίδιο και όσον αφορά τα θέματα υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή είχαμε και το Ευρωπαϊκό Έτος Αναπηρίας πριν από κάποιο διάστημα, υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ ανδρών με αναπηρία και γυναικών με αναπηρία. Αν δείτε και στο Κοινοβούλιο, ο πρώτος ε, ε, ευρωβουλευτής είναι άντρας με αναπηρία. Είμαι βέβαιη ότι η Άγγελα θα κάνει μια πολύ καλή έκθεση και στη δημόσια Κρόαση ακούσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Next is Mrs. Papadopoulou. Please, you have the floor. κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, Πράγματι έγινε μία ακρόαση την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, διότι όλοι όσοι ήμασταν εκεί παρόντες, θεωρήσαμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλά και ισορροπημένη έκθεση αυτή. Συμφωνώ με τη Ζήτα ότι οι γυναίκες με αναπηρία ε, αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση και γιατί είναι γυναίκες και γιατί είναι άτομα με αναπηρία. Ε, προβάλλονται στα μέσα μεν, αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Ορισμένες φορές είναι και ε, θύματα βίας, ακόμα και από άτομα στο στενό του οικογενειακό περιβάλλον ή από τους ανθρώπους που τους φροντίζουν και δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νέου. Θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως ίσους και ως ε, ε, φερόμαστε και στα υπόλοιπα άτομα με αναπηρία. Καταθέσαμε και σχετικές τροπολογίες, επισημέναμε το γεγονό ότι υπάρχουν και γυναίκες αλλά και νεαρά κορίτσια με αναπηρία. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και όσον αφορά τις συνέπειες ε, της οικονομικής κρίσης ε, γυναίκες και νέα κορίτσια με αναπηρία, καταθέσαμε και σχετική τροπολογία γιατί θεωρούμε ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, μέτρων λιτέτητας και περικοπών στον προπολογισμό, οι γυναίκες με αναπηρία όντω υποφέρουν διότι είναι στις πιο ευάλωτες ομάδες. Τονίσαμε επίσης ότι όλα τα ε, κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχές ε, στην παιδεία, στην κατάρτιση, στην απασχόληση και φυσικά να έχουν τις ίδιες δυνατότητες κοινωνικής ένταξης, έχουν το δικαίωμα στην εγκυμοσύνη και στη μητρότητα, ακόμα και με την αναπηρία τους, ε, χρειάζονται όμως ειδική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και επιπλέον πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη κατάρτιση όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία. Χρειάζονται ειδική κατάρτιση για να μπορούν να τους ε, ε, μιλούν, να τους ακούν και να ανταποκρίνονται στις ε, ειδικέ τους ανάγκες. Και επίσης ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους, ιδίως γυναίκες και νέα κορίτσια με αναπηρία γιατί είναι στις ευάλωτες ομάδες και πρέπει να γίνει και κατάλληλη συλλογή στοιχείων και δεδομένων για να έχουμε σχεδιασμό και των κατάλληλων πολιτικών. Και πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι είναι και στα δύο φύλλα η αναπηρία στα κράτη-μέλη. Κατά τα λοιπά να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση διότι επισημαίνει αρκετούς τομείς, περιλαμβάνει τα πάντα και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων ε, και τις συμφωνίες ε, οι οποίες άπτονται των θεμάτων αυτών, καλύπτει όλα τα θέματα και μάλιστα με πολύ καλό τρόπο. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την ε, έκθεσή της. Ε, καταθέσαμε κάποιες τροπολογίες διότι θα θέλαμε να διευκρινιστεί το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία, γιατί γίνεται η διάκριση μεταξύ των δύο και εξετάζεται και η προπτική των κοριτσιών ως μια διαφορετική προπτική. Ε, αναφερόμαστε όχι μόνο σε σωματική αναπηρία, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η πνευματική αναπηρία και κοινωνικο-κινητικές ε, ε, δυσκολίες και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο, ο όρος άτομο με ειδικές ανάγκες, διότι εδώ και καιρό έχει αντικατασταθεί από τον όρο άτομο με αναπηρία και επίσης μας ενδιαφέρουν και κάποιες ε, συνολικές δυνατότητες πρόσβασης, ε, πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, τεχνολογικές συσκευές, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην παιδεία, στην δυνατότητα γραφής, οποιαδήποτε δυνατότητα χρήσης μηχανών, ακόμα και έκδοσης εισιτηριών, ε, γυναικολογικές ε, ιατρικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις γυναίκες αυτές ε, και φυσικά και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην αρμόδια επιτροπή συζητήθηκε και το θέμα της πρόσβασης στην ψηφιακή εποχή, διότι είναι πολύ σημαντικό στην ψηφιακή εποχή να μπορούν και τα άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν ε, τις ψηφιακές δυνατότητες και κυρίως οι γυναίκες με αναπηρία. Και όχι μόνο όσον αφορά την, ε, το οπτικοακουστικό ε, υλικό αλλά και άλλες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ένα κορίτσι με σύνδρομο Down για να μπορεί να ε, έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο χρειάζεται κάποια απλή προσαρμογή. Το ίδιο νέο γραμμένο με απλό τρόπο θα είναι πολύ πιο εύκολο να το διαβάσει οποιοδήποτε άτομο με αναπηρία. Η πρόσβαση λοιπόν στο διαδίκτυο αλλά και στο περιεχόμενο του διαδικτύου ώστε τα άτομα με πνευματική αναπηρία να μπορούν να κατανοήσουν τι γράφεται, να υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία θα εξηγούν κάποια πράγματα με νοηματική γλώσσα και ζητάμε και κατάλληλη επιμόρφωση και κατάρτιση όποιου όλου των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, ώστε να μπορούν να συμπεριφερθούν με κατάλληλο τρόπο στα άτομα και στις γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία και φυσικά όσον αφορά και την ε, πνευματική διανοητική στέρηση, διότι με την ε, σωματική αναπηρία ο κόσμος δείχνει περισσότερο κατανόηση, αλλά η διανοητική και πνευματική αναπηρία αποτελεί στίγμα. Και τα δημόσια συστήματα υγείας ε, θα πρέπει να μπορούν να εντοπίσουν ε, τα άτομα αυτά τα οποία βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση και να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα ώστε να τους δίνεται ιδέουσα προσοχή. Όσον αφορά το θέμα της μητρότητας, ε, ζητήθηκε να υπάρχει μια μεγαλύτερη άδεια μητρότητα για τις γυναίκες με αναπηρία. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο διότι υπάρχουν πολύ περισσότερες προκλήσεις που δεν έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα χωρίς αναπηρίες και φυσικά ζητούμε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τη σεξουαλικότητά τους ελεύθερα, να ξεφύγουν από τις προκαταλήψει που υπάρχουν για να μπορέσουν να ζήσουν τη σεξουαλικότητά του δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι γυναίκε με αναπηρία είναι πάντα γυναίκες και θα πρέπει να σπάσουν αυτές οι προκαταλήψεις και θα μπορούν, πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ε, για την αναπαραγωγή, τον οικογενειακό προγραμματισμό και το δικαίωμα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους όπως και όλες οι υπόλοιπε γυναίκε που δεν έχουν αναπηρία. οι γυναίκες και τα νέα κορίτσια που βρίσκονται σε ίδρυμα ε, θα πρέπει να έχουν κατάλληλη φροντίδα και υπηρεσίες υγείας και γι' αυτό ακριβώς καταθέσαμε ε, τροπολογίες ώστε να μην δίνονται ποτέ αντισυλλεπτικές μέθοδες, μέθοδοι ή να μην τους προσφέρεται η άμβλωση σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία θέλει να διατηρήσει την εγκυμοσύνη. Δηλαδή ε, να μην μπορεί κανείς να αποφασίσει για την αναπηρία τους χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους. Εάν το άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να δώσει τη σύμφωνη του γνώμη, για παράδειγμα για τη στήρωση, για την άμβλωση, όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια της νομιμότητας, θα πρέπει όσον αφορά τη συγκατάθεσή του να βασιζόμαστε πάντα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε αυτή την περίπτωση τη συγκατάθεση θα πρέπει να τη δίνει ε, η οικογένεια ή ο νόμιμος κηδομόνας ή το άτομο που τους εκπροσωπεί. Ζητήσαμε επίσης και μέτρα για να εντάξουμε δείκτες σε εθνικό επίπεδο που αφορούν την προοπτική των φύλων και επίσης να δώσουμε και περισσότερα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που θα λαμβάνουν υπόψη και τη διάσταση του φύλου αλλά και τη σχέση φύλου και αναπηρίας. Και επίσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι ε, τακτικές... Ε, ε, αναφορές και εκθέσεις που θα γίνονται από πλευράς κρατών μελών θα πρέπει να περιλαμβάνουν πάντα πληροφορίες για γυναίκες και νέα κορίτσια με αναπηρία ώστε να έχουμε μια πιο ε, καλή αποτύπωση του τι ακριβώς σημαίνει ανα πάσα ε, στιγμή. Και επίσης θέλουμε και κάποια στοιχεία για τη βία, ιδίως για τα κορίτσια και πρέπει να ληφθούν και κάποια νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσουμε τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια με αναπηρία και εντός και εκτός της οικογενειακής τους αιστείας ε, και σε περίπτωση που υπάρχει κακό μεταχείριση και βία και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα άτομα αυτά με αναπηρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για να βελτιώσουμε το επίπεδο ένταξης και πρόσβασης των γυναικών και των ε, κοριτσιών, ώστε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Ξέρετε ότι στη Γενέβη, στα Ηνωμένα Έθνη, υπήρξε και μια ομάδα εργασίας στην οποία είχα την ευτυχία να συμμετέχω για να γίνει πραγματικά έκκληση προς όλες τις επιχειρήσεις και προς όλες τις ε, διοικήσεις για να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές ε, στις θέσεις εργασίας ώστε να μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να έχει πρόσβαση στις θέσεις αυτές εργασίας. Και είναι διάκριση να μην γίνονται αυτές οι προσαρμογές στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό που θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία, ιδίω οι γυναίκες με αναπηρία, γιατί είναι αντικείμενο διπλής διάκρισης, ε, διότι είναι και γυναίκες και άτομα με αναπηρία, και τα κορίτσια να είναι ισότιμες απέναντι στον νόμο και να έχουν το ίδιο δικαίωμα προστασίας ενώπιον του νόμου και να χαίρουν τον ίδιων ωφελών με όλους τους υπολείπους. Θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι το λίκνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό φυσικά θα πρέπει να μεταφράζεται σε όλες μας τις δράσεις και πραγματικά θεωρώ ότι η έκθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφορά ε, για να υλοποιήσει το όνειρο τόσων πολλών γυναικών και νέων κοριτσιών με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής, ε, σωματική, ε, ψυχική ή είναι τυφλά άτομα και φυσικά θα πρέπει να μπορούμε να πείσουμε αυτές τις κοπέλες και γυναίκες ότι όντως είναι ισότιμες απέναντι σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Γνωρίζουμε όλα αυτά τα σημεία που αναφέρατε και τα έχουμε επεξεργαστεί σε μία μελέτη η οποία ενσωματώθηκε το 2010 στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία και στις βασικές δράσεις 2010-2015 για τον τομέα αυτό. Αυτή η στρατηγική για την αντιμετώπιση της αναπηρίας περιλαμβάνει την αρχή ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε όλους αυτούς που υποφέρουν από μια αναπηρία να μπορέσουν να αναλάβουν αυτές ε, τις ε, δυνατότητες, να τους στηρίξουμε σαν ε, άτομα που θέλουν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας ή σαν φοιτητές ή σε άλλες δραστηριότητες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και βεβαίως θα πρέπει την ίδια ώρα να εφαρμόζεται στην Ευρώπη η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για άτομα με αναπηρίες. Προετοιμάζουμε επίσης τη νέα στρατηγική που θα δημοσιευθεί αργότερα το 2013. Και βεβαίως σε όλες αυτές τις δράσεις γίνεται ένα gender mainstream. Σε όλες τους τομείς της στρατηγικής για την αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε, κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο για τις συνεισφορές τους και νομίζω ότι με τις τροπολογίες η έκθεση αυτή θα εμπλουτιστεί και θα γίνει μια καλή έκθεση. Ε, ελπίζω να μπορέσω να συμπεριλάβω όλα αυτά και να τα λάβω υπόψη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω. Κύριε Βέρτμαν, σας ευχαριστούμε για τις τροπολογίες. Η προθεσμία είναι 5 η ώρα στις 15 ε, Ιουλίου. Θα συζητήσουμε 2 ή 8 Σεπτεμβρίου και θα ψηφίσουμε στις 3 Οκτωβρίου. Νομίζω τελειώσαμε με το σημείο 15 και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 16. Πρόκειται για την εκβιομηχάνηση Ευρώπης, για την ε, προώθηση ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας και θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών για μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ίτρε, Η εκ νέου βιομηχανίση της Ευρώπης πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθεί μια ισχυρή, πολύμορφη βιομηχανική βάση με, που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας ταυτόχρονα όμως και θα ε, υλοποιεί τις ευκαιρίες που θα έχει. Η ισότητα έχει ευκαιρία να δώσει λοιπόν αυτή την ανάπτυξη και θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ε, κάτι που παίζει ζωτικό ρόλο στην ε, νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Δυστυχώς έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η διάσταση του φύλου δεν έχει συμπεριληφθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής για μια πιο ισχυρή βιομηχανία για ανάπτυξη και εξυγίανση καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προωθήσουν και να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών με προγράμματα, να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ε, και επίσης να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση ε, των ε, γυναικών επιχειρηματιών σε διάφορες μορφές χρηματοδότησης, δανεισμό και επιχειρηματικά κεφάλαια. Επίσης ε, καλούμε να, τα κρατη να λάβουν όλα τα μέτρα για την ε, ανατροπή των στερεοτύπων ε, της μη συμμετοχή των γυναικών στην επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και τα μαθηματικά και να κάνει την πρόσβαση των γυναικών σε αυτές τις επιστήμες πιο εύκολη. Επίσης, Ζητάμε από τα κρατημέλη να συνδυάσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με πολιτικέ απασχόλησει για τι νέε γυναίκε για να περιοριστεί ο ρυθμό των ε, νέων γυναικών που εγκαταλείπουν ε, την ε, εκπαίδευση και Τέλος, θέλουμε να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή, η ισόρροπη συμμετοχή των ε, δύο φύλων ε, να διασφαλίζεται στις ομάδες δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αυτά συνοπτικά κύριε Πρόεδρε, δεν είχαμε και πάρα πολύ χώρο για... Είχαμε μόνο δύο σελίδες. Είχαμε λοιπόν περιορισμένο χώρο, γι' αυτό προσπάθησα να είμαι σύντομη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ε, θα καλωσορίσω όλες τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κράτσα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδοπούλου για την γνωμοδότηση αυτή που έκανε σε μια πολύ σημαντική έκθεση της Ήτρε, διότι είναι μια μεγάλη, ε, μεγάλος στόχος για την Ευρώπη να επανακτήσει τη βιομηχανική της παραγωγή και τον βιομηχανικό δυναμισμό της. Το ευρωπαϊκό θαύμα στηρίχτηκε πάνω στην βιομηχανική επανάσταση. Οι επιστήμες, η τεχνολογία, η ανάπτυξη της τεχνολογίας συνδέεται με την ιστορία της Ευρώπης και είναι κρίμα σήμερα να έχει αυτή την κρίση βιομηχανικής παραγωγής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ανακαλύπτουμε ότι εκτός από την προώθηση της καινοτομίας, ε, της ε, ε, εφαρμογής της επιστήμης ε, στη βιομηχανία. Χρειαζόμαστε και ανθρώπινο δυναμικό και, ε, και καινοτομία. Και εδώ οι γυναίκες έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό, διότι είναι ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί για το, όλους τους τομείς που μπορούν να αφορούν την, την βιομηχανία σήμερα. Και δεύτερον, είναι ένα ανθρώπινο δυναμικό με πολλές ιδέες, ταλέντα, τα οποία χρειάζεται σήμερα η βιομηχανοποίηση της Ευρώπης. Διότι πρέπει να κάνουμε σαφές και θα το κάνω, προσπαθήσω να το αναδείξω με ε, σύντομε τροπολογίε ότι η βιομηχανοποίηση της Ευρώπης έχει να κάνει με όλους τους τομείς Από τις νέες τεχνολογίες μέχρι την αναβίωση των παραδοσιακών βιομηχανιών της Ευρώπης Κάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο και με την τεχνογνωσία των γυναικών και τη δυνατότητα ε, εκπαίδευσή τους αλλά και με την ε, ε, περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό, εντάξει, δεν είμαστε Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά αυτό έχει σημασία διότι ε, με την βιομηχανοποίηση δεν συνδέονται μόνο οι γυναίκες μηχανικοί, οι γυναίκες επιστήμονες, αλλά συνδέονται και οι γυναίκες που, είναι, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις παραδοσιακές βιομηχανίες στην περιοχή τους, που έχουν σχέση με μια δεξιοτεχνία, με μια δεξιότητα την οποία οι γυναίκες ή έχουν, εύκολα μπορούν να αποκτήσουν ή να εξελίξουν. Το ότι χάνουμε την παραγωγή της πορσελάνης στην Ευρώπη, το ότι χάνουμε το τεξτάρι στην Ευρώπη. Αυτά έχουν να κάνουν με ε, παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα, τα οποία έχουμε κάθε συμφέρον να τα αναπτύξουμε και να τα διατηρήσουμε. Ε, αυτό είναι κάτι έτσι ιδιαίτερο που έχω να, σημειώσω και να προσθέσω. Όσο για την ε, ε, από την άλλη πλευρά την πρόσβαση στη, στο, στη χρηματοδότηση σε αυτά που αναφέρει η κυρία Παπαδοπούλου συμφωνώ απόλυτα οι γυναίκες μπορεί να γίνουν και επιχειρηματίες στον τομέα της, ε, ε, της βιομηχανίας και γι' αυτό χρειάζεται η υποστήριξή τους και η πρόσβασή τους στα μέσα είτε αυτά έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, είτε έχουν να κάνουν με τις ομάδες απόφασης, είτε έχουν να κάνουν με την ε, χρηματοδότηση. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές θέλω να πω, ε, που είναι πολύ σημαντικά ε, για το πολιτική μου ομάδα πώς θα αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες επαναλαμβάνω, που έχουν να κάνουν με όλους τους τομείς από τις νέες τεχνολογίες μέχρι την παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία που χάνεται σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Γιώχανσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή της πρόταση. Είμαι σκιώδης εισηγητής ε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας για την ίδια έκθεση Οπότε μπορώ να μεταφέρω εκεί πολλά από αυτά τα σχόλια που άκουσα από την εισηγήτρια. Χρειάζεται να βρεθεί κατάλληλη θέση για αυτά τα σχόλια και τις προτάσεις στην έκθεση, διότι είναι άτομα τα οποία επηρεάζονται. Μάλιστα στις... Ε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα της βιομηχανίας, έτσι ώστε όλος ο πολίτης, όλος ο πληθυσμός να μπορεί να βρει δουλειά. Πιστεύω πως η έκθεση είναι καλή, πολύ δυνατή και πρέπει να ασχοληθούμε με ορισμένα ε, οικονομικά ζητήματα τα οποία πλήττουν διαφορετικά τις γυναίκες. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα τα οποία παρέχουν κεφάλαιο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δεν είναι το ίδιο για όλους. Επίσης, ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό. Πρέπει, πιστεύω, να τονίσουμε τις δυνατότητες που έχει η διαβίου μάθηση. πολλές φορές τα αγόρια, τα κορίτσια οδηγούνται σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό δρόμο και δεν αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που έχουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εστιάσουμε και στην ε, εκπαίδευση ενηλίκων. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα κορίτσια και τα αγόρια θα έχουν την ευκαιρία να αλλάζουν κατεύθυνση αργότερα. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να αλλάξει διδρομία όταν είναι 30 ή 40 χρονών. Μπορούμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε ορισμένα από αυτά τα σημεία. Μετά, αναφέρατε και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος ανέφερε τη χώρα μου, τη Σουηδία, νωρίτερα. Και στη Σουηδία συνήθως τα αγόρια είναι αυτά τα οποία αποκλείονται από την εκπαίδευση και την απασχόληση. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές περιστάσεις ε, στην κάθε χώρα. Και επίσης ε, είναι διαφορετικό αν μεγαλώνει στην Ήπεθρο ή στην πόλη. Σημαντικό πάντως είναι και κορίτσια και αγόρια να έχουν καλή εκπαίδευση και να έχουμε εμείς την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια ε, σωστή και λειτουργική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για τη γνωμοδότηση. Συμφωνώ ότι είναι λάθος και λυπηρό ότι τα, το θέμα της ποιότητας ε, δεν λήφθη υπόψη στην έκθεση. και πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε στοχεσμένες παρεμβάσεις έτσι ώστε να ε, συμπεριλάβουμε το θέμα της ποιότητας. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή οικονομική ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία για την αύξηση της απασχόλησης και η ισότητα της απασχόλησης και η ισότητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Σίγουρα θα επικοινωνήσω μαζί σας για τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω εγώ το λόγο, διότι είμαι και εγώ σκιώδης εισηγητής το θέμα αυτό και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, πολύ καλή πρόταση. Έχουμε μια πολύ καλή αφετηρία εδώ. Τρία σημεία είναι πάρα πολύ καλά. Και τρία θα μπορούσαμε επίσης να τα επεξεργαστούμε περισσότερο. Καταρχάς πιστεύω πως είναι σημαντικό στην πρώτη παράγραφο όπου αναφέρεται η έλλειψη της ε, προοπτικής ποιότητας. Στην έκθεση κανείς δεν σκέφτηκε την ποιότητα. Πράγματι, κανείς δεν σκέφτηκε πώς αυτό επηρεάζει τους άντρες και τις γυναίκες. Επίσης, το σημείο 5 πιστεύω ότι είναι αρκετά καλό που ζητάτε από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα πετούμενα μέτρα για την ανατροπή των στερεοτύπων ότι η επιστήμη, η τεχνολογία και τα μαθηματικά είναι ανδροκρατούμενοι τομείς. Πιστεύω πως εδώ πρέπει να γίνουν πάρα πολλά και γι' αυτό είναι σημαντικό να δούμε ποια μέτρα μπορούμε να βρούμε για να χρησιμοποιήσουμε. Είναι πράγματι αληθές ότι οι άνδρες και οι γυναίκες χρειάζονται αργότερα ε, στη ζωή τους ε, πολλές φορές ε, κίνητρα για να αλλάξουν διοδρομία. Πολλές φορές τα αγόρια και τα κορίτσια μεγαλώνουν με λάθος πρότυπα που τους δίδονται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αλλάξει αυτό και να δοθούν προοπτικές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να απαλλαγούμε από τα στερεότυπα που περιορίζουν την ελευθερία του ατόμου. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ και η παράγραφος 8 όπου τονίζει ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων στον χώρο εργασίας. Τώρα, τρία σημεία πιστεύω πως θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο. τα στερεότυπα. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει μια βιομηχανική πολιτική που προωθεί τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Αυτό χρειάζεται δουλειά σε πολύ πρώιμο στάδιο, από νωρί, όταν πας δηλαδή σε ένα μαγαζί παιχνιδιών. Τώρα, βλέπουμε ότι από τη μία μεριά είναι όλα ροζ, φροντίδα, κούκλες και από την άλλη είναι όλα γαλάζια, Υπάρχουν δραστηριότητες, κατασκευαστικά παιχνίδια που τα γόρια μπορούν να χτίσουν εκεί. Είναι λοιπόν φυσικό επόμενο τα αγόρια και τα κορίτσια να ε, ακολουθούν διαφορετική πορεία. Προσωπικά εγώ αισθάνομαι ότι έχω το 50% μόνο των δυνατότητων που θα μπορούσα να έχω και όχι το 100% ως άντρας. Επίσης, ε, στο σημείο 4 έχουμε διαφορετικές απόψεις. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, μεν, αλλά όταν μιλάμε για κεφάλαια κινδύνου, εσείς ε, λέτε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετική αφετηρία. Όμως ε, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό και όχι απαραίτητα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με όσα αναφέρονται στο σημείο 4, όμως πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι τα σχολεία. Ο κύριος Γιώχανσον είναι Σουηδός και αυτός και θέλω να απαντήσω ότι στη Σκανδιναβία το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε είναι τα αγόρια. Τα αγόρια εγκαταλείπουν προώρα το σχολείο, τα αγόρια αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα εκεί. Και ακούμε πολύ συχνά ότι οι γυναίκες ε, υφίστανται διακρίσεις σε τόσους πολλούς τομείς, αλλά στη Σουηδία υπάρχει το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα. Τα αγόρια είναι αυτά που αποκλείονται και όταν διαβάζω τη διατύπωση εδώ, μου φαίνεται κάπως ότι δεν συμπεριλαμβάνεται και τα αγόρια ως ε, ακόμα μια ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή γνωμοδότηση και θα καταθέσω ορισμένε σε πολύ συγκεκριμένε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ήθελατε να σχολιάσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ όχι, τότε ε, κύριε Παπαδοπούλου έχει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση δεν ήξερα ότι στη Σουηδία έχετε πρόβλημα με τα γόρια που εγκαταλείπουν το σχολείο. Στη χώρα μου οι γυναίκες πραγματικά αριστεύουν ε, και στους μεταπτυχιακούς τίτλους ε, και είδα και μια συγκριτική μελέτη της Eurostat πρόσφατα και από ό,τι είδα οι γυναίκες βρίσκονται σε πολύ υψηλά ακαδημαϊκά επίπεδα αλλά όταν στη συνέχεια ε, του ζητείτε να ενταχθούν στη γυναική επιχειρηματικότητα. Δυστυχώς στον ε, χώρο των επιχειρήσεων είναι πολύ περισσότεροι οι άνδρες παρά οι γυναίκες. Ε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ώστε να ε, ισοσκελίσουμε την ακαδημαϊκή αριστεία με την επιχειρηματική αριστεία των γυναικών. Ε, ίσως δεν είναι πρόβλημα στη Σκανδιναβία γιατί είναι διαφορετικές οι πολιτικές ε, ε, εδώ και αρκετά χρόνια. Στις σκανδιναβικές χώρες γίνονται πολλά πράγματα σε θέματα ισότητας των φύλων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας. Πραγματικά είναι πολύτιμα όλα όσα μας είπατε και φυσικά θα τα λάβω υπόψη. Θα καταθέσω και εγώ κάποιες τροπολογίες όπως είπα, διότι όταν κάποιος ε, συντάσσει μια γνωμοδότηση είναι περιορισμένος ο χώρος και προσπαθούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα, αλλά όταν κατατίθεται τροπολογίες μπορούμε ίσως να ε, έχουμε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω λίγο το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 15 Ιουλίου 5 η ώρα το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, 15 Ιουλίου 5 η ώρα το απόγευμα και έχετε ε, δυνατότητα ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 21 Σεπτεμβρίου. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 17 Γενικός Προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 για όλα τα τμήματα. Η συντάκτηρα της γνωμοδότησης είναι η κυρία Ματέρα, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν είναι παρούσα και θα την αντικαταστήσει κάποιο συνάδελφος. Παρακαλώ, η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να αναβάλουμε το σημείο αυτό, διότι αν υπάρχει θα το προτιμούσα. διότι τα στοιχεία που μου έδωσε η κυρία Μάτερα είναι αρκετά προβληματικά. Καλύτερο θα ήταν λοιπόν να το αναβάλουμε. Εγώ βέβαια θα μπορούσα να σας πω εκ μέρους της ε, όλα όσα μου έχει στείλει, αλλά ακόμα και η πρώτη φράση δημιουργεί αμφιβολίες διότι λέει ότι το σχέδιο προπολογισμού περιλαμβάνει ελάχιστες αναφορά στην ισότητα των φύλων, δεν υπάρχει συγκεκριμένος προπολογισμός για την ε, ισότητα και δεν λαμβάνεται υπόψη ε, δεόντως η διάσταση του φύλου. Και φυσικά υπάρχουν αρκετές, αρκετά σημαντικά σημειώσεις ποσών. Θα προτιμούσα λοιπόν να είναι κάποιος εδώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ακούσει όλα όσα έχουμε να του πούμε ή αλλιώς να αναβάλουμε το συγκεκριμένο σημείο, διότι έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται και τη δική σας την παρέμβαση. Υπάρχει κάποιος από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα θέλει να απαντήσει και να πει κάτι από αυτού. Παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Το σχέδιο προπολογισμού του 2014 αντανακλά τη δομή που θα έχουμε πλέον στο νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες γραμμές προπολογισμού που φαίνονται διαφορετικά από ό,τι τις είχαμε μέχρι τώρα. Μας ενδιαφέρουν οι 330202 που περιλαμβάνει την προηγούμενη 320601 και 330602 ήταν το προηγούμενο πρόγραμμα προόδου ε, τα θέματα κατά της των διακρίσεων και το θέμα της ισότητας των φύλων. Πέραν αυτών, η άλλη σημαντική ε, γραμμή ε, προπολογισμού είναι η 320201 που περιλάμβανε τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το πρόγραμμα για την ε, υπηκότητα και είναι αλήθεια ότι ε, έχουν αλλάξει οι αριθμοί στις γραμμές προϋπολογισμού και δεν αντανακλούν τη μεταφορά από την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο στην παρούσα, αλλά τα ποσά μεταξύ των προηγούμενων και των τρεχουσών ε, ποσών είναι λίγο πολύ τα ίδια. Διατηρούμε αντίστοιχο προϋπολογισμό και αντίστοιχα ποσά και συνάδουν με αυτά τα οποία είχαμε προβλέψει για τον προϋπολογισμό του 2014. Η κυρία Μπάουερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε αυτά που μου έχει να μας πει η κυρία Ματέρα. Δυστυχώς ε, είναι ασθενής και στελεμένα στη θέση της λέει ότι το σχέδιο προπολογισμού περιλαμβάνει καταρχήν ελάχιστε αναφορέ στην ισότητα των φύλων, όπω είπα προηγουμένω, και η διάσταση του φύλου με εξαίρεση τον τίτλο 21 βρίσκεται στο σημείο 08 επίσης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη να ενισχύσουμε την ε, ε, συμμετοχή και το ρόλο των γυναικών ε, στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Αυτό έχει αφαιρεθεί και υπάρχουν και άλλα σημεία, κάποιες άλλες γραμμές προπολογισμού, για παράδειγμα η 150301 που έχουμε διάφορους υπολογισμούς εκεί, η γέννηση νέων δεξιοτήτων και καινοτομία, καμία αναφορά στη διάσταση του φύλου, επίσης και στο πρόγραμμα για τις κοινωνικές αλλαγές και τις καινοτομίες, καμία αναφορά στη διάσταση του φύλου. Δεύτερον, σε αρκετές περιπτώσεις ε, το επίπεδο των ε, δεσμεύσεων υποχρεώσεων σε σχέση με τις ε, πληρωμές έχει μεγάλες διαφορές. Για παράδειγμα, η 330201, η γραμμή προπολογισμού για να διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων και την ενδυνάμωση των πολιτών, η 030202 που προάγει την έλλειψη διακρίσεων και την ε, ισότητα ε, έτυχε μια πολύ προσεκτικής προσέγγισης ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2013 και τη λιτότητα. Εδώ τίθεται ερωτηματικό και δεύτερον, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη βία κατά των γυναικών. Είναι συγκεκριμένο στόχο τη 330201 για να διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων και την ενδυνάμωση των πολιτών. Εκεί δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στον τίτλο, αλλά ούτε στις παρατηρήσεις. Η συγκεκριμένη γραμμή προϋπολογισμού έχει ε, και τους πόρους για την παρακολούθηση του προγράμματος Δάφνη και το θέμα της ηθαγένειας. Το θέμα είναι πού θα τα βρούμε αυτά τα κονδύλια. Ίσως η εξήγηση είναι ότι ο προγραμματισμός έγινε επί τη βάση της παρούσας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχει λάβει υπόψη τις διαπραγματεύσεις τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα προγράμματα περιθαγένειας ε, υποτίθεται ότι θα παρακολουθούσαν αρκετά προγράμματα συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος Δάφνη. Επομένως, μία αναφορά ε, στη βία κατά των γυναικών κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον στις παρατηρήσεις. Υπάρχει και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δεσμεύσεων πληρωμών για την ε, ολοκλήρωση των ε, θεμάτων ηθαγένειας στη γραμμη 56.5.2.1.3.1 το 2013 σε σχέση με τη 41-33-00 το 2014. Ποια είναι ο λόγος για αυτή τη διαφορά. Και επίσης, ε, οι δαπάνες για τα δικαιώματα των πολιτών, υπάρχει μία μίεση που είναι άνω του 15% σε αυτή την περίπτωση. και σε δεσμεύσεις ε, υποχρεώσεων και σε δεσμεύσεις ε, πληρωμών. Ποιος είναι ο λόγος. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις εξελίξεις, Δεν θα ήθελα να σας επιβαρύνω και με ένα ακόμα καθήκον, αλλά νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι καλό θα ήταν να στείλουμε μια επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, διότι έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπάουερ. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέσσερα πράγματα νομίζω είπατε. Καταρχάς είπατε ότι υπάρχει ελάχιστη αναφορά στο θέμα της ισότητας των φύλων. Δεύτερον, το επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων ε, και των πληρωμών έχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές εδώ και όπως είπε και η κυρία Μπάουερ δεν ξέρω ε, αν αυτό δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο. Το γεγονός ίσως ότι κάποια προγράμματα θα αρχίσουν να ισχύουν στα τέλη του 2013 και στη λιτότητα ε, και επίσης ε, λέγεται ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη βία κατά των γυναικών και γνωρίζετε ότι η Επιτροπή μας πραγματικά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα Δάφνη με τον, είδε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο είτε στη συγκεκριμένη γραμμή προϋπολογισμού είτε οπουδήποτε αλλού και επίσης βλέπουμε μεγάλη διαφορά ε, για τα, ε, ο προϋπολογισμό, τη γραμμή για τα δικαιώματα των πολιτών. Μπορείτε να μας απαντήσετε κάτι τώρα, θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερος. So, as κυρία Ο προϋπολογισμός, κυρίως για το πρόγραμμα, βασίστηκε στην πρόταση της Επιτροπής του 2011. Δηλαδή, όπως αναπτύχθηκαν στις διαπραγματεύσεις και δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στο έγγραφο αυτό. Και όσον αφορά τα προγράμματα, μπορώ να σας δώσω επιπλέον επεξηγήσεις. Γίνονται πολλές αναφορές και στη βία κατά των γυναικών και στην ισότητα. Δεν υπάρχουν όμως αυτό το έγγραφο γιατί δεν υπήρχαν το 2011 στις προτάσεις της Επιτροπής. Το 2015 θα βασιστούμε στην υιοθέτηση του προγράμματος και φυσικά Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να ενσωματωθούν και οι αναφορές στα προγράμματα για τη βία κατά των γυναικών, την ισότητα των φύλων και το gender mainstreaming. Δυστυχώς δεν φαίνονται αυτά αυτή τη στιγμή στο έγγραφο, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι βασιστήκαμε στις προτάσεις, επαναλαμβάνω, του 2011. Θα συνεχίσει ο συνάδελφος. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά όσον αφορά τις πιστώσεις δεσμένων και τις πιστώσεις πληρωμών, θα πρέπει να καταλάβετε ότι η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται για τις ε, πιστώσεις δεσμεύσεων στην συμφωνία του 11 η οποία τελικά οδήγησε σε μείωση των ποσών κατά 16,6 στο τμήμα 3. Αλλά πρόκειται για δεσμεύσεις που αν δείτε το ποσό τους αντιστοιχεί ακριβώς αυτό που φαίνεται σήμερα στο έγγραφο. Τώρα, όσον αφορά τις πληρωμές, όντως υπάρχει διαφορά με τις δεσμεύσεις. Και βεβαίως πρόκειται για το πρώτο έτος υλοποίησης των προγραμμάτων και μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε αυτήν την επιφυλακτική και προσεκτική στάση. Αυτά. Could I you, Mrs. Uh, Θέλετε να στείλουμε επιστολή? <coughs> Στον κύριο Λαμασούρ. Ναι. Νομίζω νομίζω ότι εσείς θα έπρεπε να συζητήσετε, να έρθετε σε επαφή με την κυρία Ματέρα, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι αυτά τα προγράμματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα Δάφνη θα διατηρηθούν, θα συνεχιστούν με τον νέο προπολογισμό. Πρόεδρος, δηλαδή, αν η κυρία Ματέρα και εγώ υπογράψουμε μια επιστολή, και μπορούμε εξ ονόματος της Επιτροπής να το στείλουμε, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Γίνεται αυτό. I don't know if Mrs. Matera... Δεν ξέρω αν η κυρία Ματέρα είναι διαθέσιμη, θα προσπαθήσω πάντως. Να στείλουμε μία επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμού, τον κύριο Λαμασόρ. Ωραία. Συμφωνείτε όλοι. Εντάξει. σε ευχαριστώ. Για τις τροπολογίες η προθεσμία είναι... Εδώ λέει 24 Ιουλίου. Και εγώ είχα προγραμματίσει διακοπές 24 Ιουλίου. 24 Ιουλίου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε 2 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου αν όχι 2 και 2 ή 3 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε. 18, σημείο 18, η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 2 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας. Πολύ νωρίτερα, είμαι πολύ ευτυχής. Οπότε και οι διερμηνείς μπορεί να φύγουν. Καμιά φορά αργούμε. Εδώ όμως έχουμε 50 λεπτά για τους διερμηνείς. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Ευχαριστώ την γραμματεία. Ευχαριστώ πολύ όλους τους διερμηνείς που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε μέν τους δε και να επικοινωνήσουμε. Και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.